Chers collègues, la séance est reprise et nous ouvrons sur un. Ξεκινάμε λοιπόν με μια ανακοίνωση της κυρίας Γκουάρδια για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε αποφασίσει πρόσφατα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς είμαστε σε ετήσια βάση αυτή μέχρι τώρα που κάναμε γνωμοδοτήσεις στην κύρια έκθεση, αλλά του χρόνου με το σύστημα της εναλλαγής θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την έκθεση. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να καταθέσουμε κάποιες συγκεκριμένες ε, ιδέες και σε αριθμό. Ε, εμείς θεωρούμε ότι η Τράπεζα των Επενδύσεων πρέπει να συμμετέχει όλο και περισσότερο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εμείς προσπαθούμε σε μόνιμη βάση να διευρύνουμε τα χρηματοδοτικά μέσα και θα θέλαμε η συγκεκριμένη τράπεζα να έχει μεγαλύτερη παρουσία. Είναι περίπλοκο το σύστημα αυτό. Ε, βέβαια, Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται τον τελευταίο καιρό. Εμείς απαιτούμε από την τράπεζα περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη ευκρίνεια. Αυτό όχι μόνο για μας συγκεκριμένα, αλλά κυρίως ε, και για τους ίδιους τους πολίτες αυτούς οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων. Απαιτείται να υπάρξει μια σύμπτωση χρονική και μια σύμπτωση θεματολογική των δραστηριοτήτων της ε, ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας αυτής και για τις επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα πρέπει κυρίως να υπάρξει συντονισμός και με την εντολή την οποία έχει η τράπεζα αυτή σε σχέση με τις επενδύσεις προς το εξωτερικό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες με τους οποίους διεξάγεται η δραστηριότητα της τράπεζας και θα πρέπει να είμαστε σε θέση και εμείς να συνεργαζόμαστε με συντονισμένο τρόπο. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να έχει μια σωστή επιλεκτική αλλά δίκαιη πολιτική. Να λαμβάνει υπόψη την σωστή διακυβέρνηση, μια σωστή λοιπόν εξωτερική στρατηγική, κάτι το οποίο αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει σαν παράδειγμα οι συνεργασίες ε, ενδιαμέσων, ε, διαμεσολαβητών, οικονομικών ενοτήτων που δεν έχουν πάρα πολύ καλή φήμη. Η καλή βαθμολογία δεν θα πρέπει να συνεργάζεται μαζί τους. Απαιτείται λοιπόν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα διαφάνεια για όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, <clears throat> οι απόψει σας θα είναι πολύτιμε για την γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ κυρία <clears throat> Γουαδιαζαβάλ ε, για τις τέσσερις ιδέες που εκφράσατε. Η κυρία Γιατεμάκη έχει ζητήσει το λόγο. Kiitoksia. <clears throat> να τα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι επιτέλους που σα βλέπω και πάλι όλου μετά τι θερινές διακοπές. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Και εκτιμώ ιδιαίτερως τα όσα μας ε, είπατε. Και συμφωνώ με τη γενικότερη γραμμή την οποία παρουσιάσατε. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου κάποια σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι συνεπή ε, στις δράσεις της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει μέτρα για να καταπολεμήσει τους φορολογικούς παραδείσους και για να καταστήσει την λειτουργία τους και την ύπαρξή τους την ίδια πιο δύσκολη, πιο δυσχερή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι είναι μάλλον κάπως περίεργο, τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί δράσεις και οντότητες οι οποίες συνδέονται με φορολογικούς παραδείσους. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως φαινόμενο. Και αυτό ασφαλώς και ανησυχεί και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Προφανώς και υπάρχουν α, ε, α, ε, σαφώς επιχειρήματα πολιτικά και νομικά που επιτάσσουν την ανάληψη δράση στο σημείο αυτό. Ένα άλλο σημείο το οποίο έθιξε η κυρία Γκάρτια Σαμπάλ, είναι το θέμα της διαφάνειας. Οι κανόνες για τη διαφάνεια και οι συνθήκες οι οποίες άλλωστε δεσμεύουν όλα τα θεσμικά όργανα προαπαιτούν διακυβέρνηση σωστή, χρηστή και διαφάνεια ε, από, όλες, ε, από όλα τα θεσμικά όργανα. Και αυτό θεωρώ ότι ασφαλώς και περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό μου φαίνεται μάλλον περίεργο που η Ευρωπαϊκή Τραπεζα, ε, Επενδυτική Τράπεζα άλλαξε το περασμένο φθινόπωρο τους κανόνες περί διαφάνειας. Και πλέον μπορεί να χαρακτηρίζει ως απόρριτα όλο και πιο πολλά έγγραφα. Αυτό αντίκειται ασφαλώς με το πνεύμα της διαφάνειας. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επίσης επεσήμενε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά το παρελθόν δεν ε, σεβόταν πάντα τους ίδιους της τους κανόνες για την διαφάνεια. Αυτό προφανώς και θα πρέπει να διορθωθεί δεδομένου και του ολοένα και μεγαλύτερου ρόλου που διαδραματίζει και τον όλο ένα και μεγαλύτερων πόρων που διατίθεται προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά γίνονται σεβαστοί οι κανόνε και έτσι δεν θα υπάρχει καμία σύνδεση προ φορολογικού παραδείσου. Αυτά από πλευρά μου. Αυτό είναι ένα ωραίο σχέδιο, η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και της ε, φορολογικής βελτιστοποίησης. Όμως αυτό υπάρχει γιατί τα κράτη-μέλη είναι αρκετά ανόητα έτσι ώστε να μπαίνουν σε φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ τους και γι' αυτό οι εταιρείε τελικά πάνε ε, και προσπαθούν να βρουν το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Αυτό τον ανταγωνισμό, τον ανόητο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να ε, τελειώσουμε και να διακόψουμε. Ποιος θα ήθελε να σχολιάσει τα λόγια της κυρίας Καρτιά Θαμπάλ. Παρακαλώ. Κύριε Μουρεσάν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την προηγούμενη ομιλήτρια. Βλέπουμε σήμερα ότι τα χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και πιο πολλαπλά και γι' αυτό χρειάζεται συνολική προσέγγιση. Σε σχέση με το ΕΦΣΥ έχει αυξηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για όλα τα κράτη-μέλη Παρ' όλα αυτά παραμένουν οι διαφορές. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διαφέρει από το ένα κράτος στο άλλο, το ε, πόσο είναι παρούσα δηλαδή. Και πρέπει να αξιολογήσουμε τις αιτίες. Υπάρχουν χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένες χρηματαγορές και χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου τα ΣΔΙΤΑ δεν είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στη διάθεσή τους. Υπάρχει έλλειμμα εκεί. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βοηθήσει όλα τα κρατημέλη να τα στηρίζει με πληροφορίε, με πυρογνωμοσύνη, με ό,τι χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά τη εργαλεία. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει γεωγραφική συγκέντρωση το καλύτερο project είναι αυτό που θα πρέπει να χρηματοδοτείται ε, και ένα παιχνίδι επί ίσης να γίνεται και αυτό δεν εφίσταται αυτή τη στιγμή. Μερικές φορές οι χώρες δεν έχουν την απαραίτητη νομοθεσία για τα ΣΔΙΤ ε, ή για άλλου τους εργαλεία και τελικά αυτό τις υπονομεύει. Υπονομεύει τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοδότησης έργων δηλαδή και θα πρέπει να προβληματιστούμε και να το διευκρινίσουμε σε συνεργασία με την τράπεζα. Η πρωτοβουλία ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και το κέντρο της Ευρώπης ήταν σημαντική, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερως με την Ανατολική Ευρώπη και σε όλες τις εκθέσεις των προηγούμενων ετών ε, το Κοινοβούλιο έχει πει ότι η πολιτική ανατολικής γειτονίας είναι πολύ σημαντική για μας ε, εν ώψη των εξελίξεων στην Ουκρανία και αλλού πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη σε όλες αυτές τις χώρες και Ε, η σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχε περιοριστεί μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια και αλλού. Θα πρέπει να περιλάβει και την Ανατολική Ευρώπη. Κατά τα λοιπά, καλωσορίζω τον ρόλο που θέλει να παίξει η Επιτροπή μας να παρακολουθήσει ε, τη δράση της ΕΤΕΠ. Ε, πολεμήσαμε σκληρά με την Επιτροπή ΕΚΟΝ και άλλες για να το καταφέρουμε αυτό και ο, ο Πρόεδρος είχε σημαντικό ε, μέρος ε, της δουλειάς αναλάβει και έτσι η Επιτροπή Προϋπολογισμών στο μέλλον θα παρακολουθήσει πιο στενά τις δράσεις Ευρωπαϊκής Τραπεζής Επενδύσεων το οποίο είναι και το σωστό να γίνει και καλώ το πετύχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρο. εάν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται να παίξει όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει προτάσει για τη δημιουργία νέου ταμείου στρατηγικών επενδύσεων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ενδεχομένω και στην Αφρική. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία και να μην επιτηρεί όλες αυτές τις δράσεις η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μόνο, να παραμείνει ε, εργαλείο της πολιτικής που μπορεί να ασκηθεί. Η κυρία Κάρτια Θαμπάλ για να ολοκληρώσει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην ίδια πλευρά, θα περιμένω τις τροπολογίες και θα παρουσιάσουμε τη γνωμοδότηση των δυνατόν συντομότερα, νωρίτερα. Ο Πρόεδρος. Καλώς καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 20 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και στη συνέχεια η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ασχοληθεί με το θέμα στις 10 ή στις 12 Οκτωβρίου. Και η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ε, ασχοληθεί με το θέμα στις 28 Νοεμβρίου και ε, το κείμενο θα εγκριθεί από την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Εάν όλα πάνε καλά. Κυρία Γκάρδια, Γκάρθια Θαμπάλ, είστε συνεισηγήτρια. Μπορείτε να πάρετε ξανά το λόγο και να μιλήσετε για την εξωτερική συνεργασία, για τα διάφορα μέσα και να πείτε τη γνώμη σας για την έκθεση της Επιτροπής για την πλατφόρμα EUBEC, την πλατφόρμα της Ένωσης. Ε, μεικτή χρηματοδότηση για την εξωτερική συνεργασία, έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες αυτής της πλατφόρμας, EUBEC. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει πράγματι να μας μιλήσει για την ε, πλατφόρμα αυτή και για τις προτάσεις που έχει. Φέτος λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό από τότε που η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεση για αυτό το πιθανό σχέδιο το επενδυτικό είναι πολύ πιο εφικτό σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει ε, τι, ποιο είναι αυτό το σχέδιο για το εξωτερικό εύση, για το επενδυτικό σχέδιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το σημαντικό είναι να ακούσουμε από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα στοιχεία για αυτό το σχέδιο, το επενδυτικό. Ο Πρόεδρος. Καλώς. Ε, θα διαβιβάσω την επιθυμία σας στον κύριο Μπρέζα και στρέφομαι προς αυτόν. Να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόεδρε. Ο κύριος Χωσέ Πες κύριος Κάιζερ από την ε, Γενική Διεθνή Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δεδομένη της ε, τη ε, ε έκθεση ε, για την περιγραφή των δραστηριοτήτων από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος 2015 και δεδομένου ότι προφανώς υπάρχει επιθυμία να εξεταστούν και οι πρόσφατες εξελίξεις στο επενδυτικό σχέδιο, θα σα παρουσιάσω καταρχάς ε, προκαταρτικά την έκθεση και θα έρθει και ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΑ σε λίγο και ο άλλος συνέδελφες θα σας παρουσιάσει το παιδιτικό πρόγραμμα λίγο αργότερα. Προκαταρτικά και από πλευρά χρονοδιαγράμματο, μια και η έκθεση δεν εγκρίθηκε ακόμα για την τρέχουσα περίοδο. Να σα εξηγήσω λοιπόν πώ έχει το ιστορικό υπόβαθρο. Θα θυμάστε πιο πολύ εξημών ότι η πρώτη εκδοχή τη έκθεση αυτή ήταν η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ε, εξωτερική συνεργασία. και συστάθηκε λοιπόν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων το 2012 μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πρώτη τέτοια έκθεση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του περασμένου έτου και παρουσιάστηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα το θυμάστε ίσω μερικοί αξιμών. σε ό,τι αφορά τη σύσταση μια τέτοια πλατφόρμα για την ε, συνεργασία, για την εξωτερική συνεργασία είχε ως σκοπό την ε, βελτιστοποίηση των επιδοτήσεων στον τομέα της εξωτερικής δράσης και προφανώς αυτή την εργασία ακολούθησαν και οι εμπειρογνώμονες από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, όπως σας είπα και προηγουμένως. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα πολιτικής που προεδρεύει τις οποίε προεδρεύει η Επιτροπή. Συμμετέχουν μέλη, τα κρατημέλη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τεχνικοί παρατηρητές και ούτω καθεξής. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη γραμματεία για την επικοινωνία και τον συντονισμό. Τέσσερι φορέ συναντήθηκε η ομάδα πολιτικής 17 ε, Δεκεμβρίου, τον 14, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2015. Τέσσερις συναντήσεις λοιπόν την προετοιμασία την είχαν κάνει οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, εκπρόσωποι τη Υπηρεσία Εκτορική Δράση, εμπειρογνώμονε και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση λοιπόν καταρχά των επενδύσεων των ιδιωτικών επενδυτών, για την αντιμετώπιση τη αλλαγή του κλίματο και το καθεξή. Και για κάθε θέμα ακολουθήσα και μια τεχνική συνάντηση. Μια τεχνική συνάντηση επίση διοργανώθηκε για την τεχνική χρηματοδότηση το καλοκαίρι του 2015. Και έτσι λοιπόν η έκθεση παρέχει μια ενημέρωση για τα θέματα τα αρθρωτικά σε ό,τι αφορά το UBEC όπως ε, ονομάζεται, θέματα διακυβέρνησης, τα μέτρα για την ε, αντιμετώπιση και την ακολούθηση των συστάσεων του Εθνικού Συνέδριου του 2014 και τη συμμετοχή και των άλλων εμπλεκομένων φορέων. Και έτσι λοιπόν ε, περιλαμβάνονται στην έκθεση και οι συζητήσει για τα ζητήματα αυτά, την καταπολέμηση του κλίματος, τη αλλαγή του κλίματος και τα βασικά πορίσματα τα οποία εξαγάγονται είναι ότι οι υπηρεσίε αυτές συνεχίζουν να δρουν αποτελεσματικά. Χρειάζεται ε, μια σαφή διακυβέρνηση. Αυτό έχει οριστεί άλλωστε και στην πρώτη έκθεση, στην πρώτη προγραμματική περίοδο. Οι πιο πολλές συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά Τα πιο πολλέ συστάσεις λοιπόν του ελεκτικού συνεδρίου λεφτήσαν υπόψη σε ό,τι αφορά τώρα το μελλοντικό έργο. Θα συνεχίσουν να γίνονται ε, συναντήσεις και μετά το Δεκέμβριο 2015 για τα βασικά ζητήματα που αφορούν το ΓΙΜΠΕΚ, δηλαδή πέρα από την προγραμματική περίοδο που ορίζεται και στην πράξη, όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, αυτό καταρχάς ήταν ε, προς απάντηση στην ε, κρίση τη μεταναστευτική του 2015. Θα το θίξει αυτό και ο συνάδελφο, αλλά εστιαζόμαστε και στι αναληφθήσεις υποχρεώσει και δεσμεύσει, και έτσι σε ό,τι αφορά τις ανάμεικτες ε, αυτές χρηματοδοτήσεις προγραμματίζονται και άλλε δραστηριότητε. Τώρα, σε ό,τι αφορά ενδεχόμενε ερωτήσει που έχετε για την έκθεση UBEC που καλύπτουν λοιπόν την περίοδο μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, α ακούσουμε πρώτα τι ερωτήσει αυτέ για να δώσουμε και την ευκαιρία στον συνάδελφο να προετοιμαστεί και να συνεχίσει μετά με την επόμενη έκθεση. Ευχαριστούμε. Έχετε ερωτήσεις, κυρία Καρτία Σαμπάλη, σε ό,τι αφορά την περίοδο Ιούλιο του 2014 μέχρι α, Δεκέμβριο του 2015. Όχι. Μάλιστα. Ο συνάδελφο σα, λοιπόν, αγαπητέ κύριε, μπορεί να πάρει το λόγο για να συνεχίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον διευθυντή μου που θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άλλες συνεδριάσεις που έχουν σχέση με την προετοιμασία του εξωτερικού επενδυτικού προγράμματος. Βρισκόμεθα υποπίεση αυτή την εποχή, γίνεται πάρα πολύ δουλειά, μας περιμένει επίσης πάρα πολύ δουλειά και γι' αυτό θα είμαι ε, συνοπτικός. Θα σας δώσω ένα, θα έλεγα, συνοπτικό, όπως είπα, σύνολο των ε, δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξεταστούν από την επερχόμενη επιτροπολογία και που θα ελεγχθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειδικότερα θα ήθελα να τονίσω ότι στα πλαίσιο της πλατφόρμας είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη πέμπτη, τρίτη συγγνώμη, την προηγούμενη τρίτη, πήραν μέρος τα κράτη-μέλη, οι χρηματοδοτικές ε, ε, υπηρεσίες, όπως σας εξήγησε άλλωστε και ο προηγούμενος συνάδελφος, σε όλους αυτούς τους εμπλεκομένους του προγράμματος επενδύσεων περιγράψαμε τις βασικές του γραμμές. Όπως επίσης γνωρίζετε, αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα είναι τμήμα της νέας εταιρικής ε, συμφωνίας πλαισίου με τις τρίτες χώρες για τα θέματα της μετανάστευσης. Είναι ένα από τα βασικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά αυτής της συμφωνίας ο βασικός στόχος αυτού του νέου ε, προγράμματος, το οποίο βασίζεται ε, θα έλεγα στην ίδια λογική όπως και το ΕΦΣΥ, το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων. Έχει τον ίδιο αριθμό πυλώνων με το προηγούμενο και συγκεντρώνει την δραστηριότητά του κυρίως στην καταπολέμηση των ε, προβλημάτων που οδηγούν στην μετανάστευση. Βασικός μας στόχος είναι να προωθήσουμε λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που γεννούν τη μετανάστευση και να βοηθήσουμε τους τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης που ε, όταν δεν υπάρχει γεννά τη μετανάστευση. Όπως είπα αυτό το επενδυτικό ε, πρόγραμμα έχει τρεις πυλώνες όπως και το FC. Ο πρώτος πυλώνας ασχολείται κυρίως με τις εμπειρίες τις οποίες αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια για τα μεικτά χρηματοδοτικά σχήματα. Αυτά τα blending facilities ε, χρησιμοποιεί αν θέλετε ε, και τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα, όπως επίσης και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και μία μορφή εγγυήσης για χρηματοδοτήσεις σε περιοχές όπου οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο πρώτος αυτός πυλώνας λοιπόν θα οδηγήσει όπως είπα στην ανάγκη δημιουργίας στήριξης ενός ταμείου εγγυήσεων, θα υποστηριχθεί από δύο άλλους πυλώνες, πρώτον τον πυλώνα της τεχνικής ε, αρρωγής, της τεχνικής βοήθειας, η οποία θα παρέχεται και στα χρηματοδοτικά όργανα, τα τοπικά αλλά και τα εθνικά, έτσι ώστε να καταστήσουμε τα όργανα αυτά ικανά να προετοιμάζουν σωστά τα προγράμματα που απαιτούνται. Τρίτον, και αυτό θα βασιστεί στις εμπειρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχουμε άλλον ένα πυλώνα, ο οποίος θα προωθήσει ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον από τις χώρες εταίρους. Βασικός στόχος προς το παρόν αυτού του προγράμματος είναι να υπάρξει ένα ενιαίο πακέτο το οποίο θα καλύψει τις επενδύσεις, τις ανάγκες των επενδύσεων στην Αφρική, στην περιοχή γειτονίας και όπως είπα και στην αρχή, το πιο σημαντικό από τα θέματα που έχουμε μπροστά μας είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα επενδυτικά σχήματα τα οποία ρευστοποιήθηκαν πρόσφατα και για την Αφρική και για την περιοχή γειτονίας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της μετανάστευσης. Πολλές χώρες στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη Τρίτη, αυτό δεν ε, φάνηκε ότι δεν θα αλλάξουμε ιδιαίτερα από αυτά που κάναμε στο παρελθόν. Με αυτά τα blending facilities εμείς στηρίξαμε κάποιους τομείς όπως οι εξηγιάνσεις, ε, των διαφόρων περιοχών, των ποαστικών ιστών, μεταφορές κτλ. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τονίσουμε τις ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα που θα μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Στο παρελθόν τέτοιου είδους προγράμματα α, ε, αντιστοιχούσαν σε ένα πολύ μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων των blending facilities που είχαμε. 5 ή 10% το πολύ. Ε, βασικός μας στόχος λοιπόν είναι να αλλάξουμε αυτές τις επενδυτικές, ε, ε, τα επενδυτικά αυτά εργαλεία, να τα καταστήσουμε πλατφόρμες που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας όμως και αυτό το, την εγγύηση για το Ταμείο της Αϊφόρου Ανάπτυξης που θα διευρύνει τις ικανότητες των χρηματοδοτικών οργάνων στον τομέα αυτό. Η διαχείριση τώρα μια τέτοια πρωτοβουλίας θα απαιτήσει μια καλύτερη συνοχή αυτό το οποίο κάνουμε σε μία περιφέρεια σαν παράδειγμα θα πρέπει να συστηματοποιηθεί για το σύνολο της Αφρικής ή για το σύνολο της περιοχής γειτονίας και θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχες δομές όπως αυτές που είχαμε κάποτε. Θα έχουμε ένα στρατηγικό συμβούλιο, το Strategic Board, το οποίο θα δίνει τις κατευθύνσεις για τη λειτουργία του προγράμματος και μετά θα έχουμε ε, συμβούλια λειτουργίας, διευθυντικά συμβούλια, τα οποία θα ασχολούνται με τη διαχείριση. Θα σταματήσω εδώ κάνοντας μία αναφορά στα ποσά. Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει ως Επιτροπή. Τα ποσά τα οποία είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση <clears throat> έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά 3,1 δις μέχρι το 20. Αυτά τα ποσά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για τη μετανάστευση συντίθενται τα ποσά αυτά 2 εκατομμύρια, 2 δι συγγνώμη το EDF, 400 εκατομμύρια από, το, από τους φακέλους του αποθεματικού, ένα δις από το DNI, επενδυτικό μέσο για τη γειτονία και 160 εκατομμύρια θα προέλθουν από το μέσο για την Αφρική ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσουμε να μοχλεύσουμε συνολικά 31 δις. 1 προς 10 η μόχλευση στην οποία προσβλέπουμε. Είναι κάτι το ε, λίγο σε σχέση με το τι πετύχαμε στο παρελθόν, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να είμαστε μετριόφρονες. Ζητάμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν τα ταμεία αυτά έτσι ώστε να υπάρξει μια συνολικότερα υψηλότερη μόχλευση από αυτήν που είχαμε μέχρι τώρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή του μηχανισμού αυτού. Ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει η μόχλευση και τα κράτη-μέλη θα ανταποκριθούν στις ε, επιθυμίες και ίσως ε, να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας και σε δημοσιονομικό επίπεδο τις ανάγκες. Λοιπόν, η κυρία Ζάμπαλ να κλείσει. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση θα ήθελα να θέσω. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μιλήσατε, αναφερθήκατε στα αριθμητικά στοιχεία που ενδιαφέρουν την Επιτροπή των Προπολογισμών, γιατί βλέπουμε το μέγεθος του θέματος, την τάξη μεγέθους και το από πού θα προκύψουν οι πόροι. Αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν σε αυτό το ταμείο. Όμως η συμβολή τους και η συνεισφορά τους θα είναι εθελοντική, θα υπάρχει μια ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά ή θα γίνει όπως έγινε και με το ΕΦΣΥ ότι τελικά νομίζαμε ότι στην αρχή όλοι θα έβαζαν αλλά τελικά έχουμε εθνική συνεισφόρα σε κοινό κορβανά. Ποιος θα τα διαχειρίζεται αυτά. Θα παραχωρηθεί η διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ακολουθηθεί κάποιο άλλο σχήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το διαχειριστεί. Πώς ακριβώς θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην μας πάρουν προνόμια και δικαιώματα για άλλη μια φορά. Μπορείτε να απαντήσετε Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. ευχαριστώ Καταρχάς, Εθελοντικέ θα είναι οι συνεισφορές που θα ζητηθούν από τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει υποχρεωτική δέσμευση μέχρι στιγμής. Οφείλω να σας πω ότι ορισμένα κράτη-μέλη στη συνεδρίαση της Πέμπτης ε, εξέφρασαν την επιθυμία να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν σε αυτή την πλατφόρμα είναι το δύσκολο κομμάτι του προγράμματος. Προφανώς θα προσπαθήσουμε όλοι να συνεργαστούν μαζί μας. Τώρα, όσο περισσότερο εφαρμόζεται και όσο πιο πολύ έρχονται τα αποτελέσματα, τόσο θα ανοίξει και η όρεξη των κρατών μελών για να συνεργαστούν για το πρόγραμμα αυτό. Τώρα, ε, ως προς τη διαχείριση, δεν το έχουμε αποφασίσει. Τα κονδυλία που χρειάζονται είναι τα εφιστάμενα. Δεν θα ζητήσουμε επιπρόσθετα. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, πολύ σημαντικό μάλιστα, γιατί ήδη είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 30% των διευκολύνσεων νέων χρηματοδότησης. Επομένως, σίγουρα θα έχει λόγο και στη διαχείριση της πλατφόρμας αυτής. Έχουν και τεχνογνωσία. Όλα αυτά θα τα αξιοποιήσουμε. Θέλω όμως να καθησυχάσω την Προεδρία, τον Πρόεδρό σας, θα είναι επαρκώς ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξη και την πρόοδο αυτού του έργου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Καλώς. Αυτά με αυτό το θέμα. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Βλέπουμε τους γενικούς προσανατολισμούς της. Προτείνω τώρα να περάσουμε στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Σαρβάμα θα πάρει το λόγο και θα μας πει πώς η Microsoft μπορεί να ανακτήσει κάποια χρήματα. Ευχαριστώ. Πράγματι, εδώ έχουμε μία άλλη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και είναι μάλιστα μία υπόθεση αρκετά μεγάλη, αρκετά μεγάλο μεγέθους που επηρεάζει 1.441 στοχευμένους δικαιούχους από τους 2.000 εργαζόμενους που απολύθηκαν στην Φιλανδία. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση παγκοσμιοποίηση. Θα θυμάστε ότι την πρώτη δεκαετία του 2000 η Νόκια κατέρευσε, την πρώτη δεκαετία ε, ήταν μάλλον ακόμα παρούσα στη δεύτερη δεκαετία όμως κατάλυσε την αγορά ε, το σύστημα Android και το λειτουργικό σύστημα της Apple. Η αίτηση όλων αυτών των ανθρώπων πληρεί τα κριτήρια που έχουν οριστεί 8,94 εκατομμύρια ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός και η συνεισφορά FG είναι 60%, 5, ε, κάτι εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Μιλούμε για απολύσεις εργαζομένων με πολλά και διαφορετικά προσόντα. Είχαμε και χαμηλών προσόντων ε, απολυμένους αλλά και υψηλών προσόντων απολυμένους. Και από τη στιγμή που είναι μια πολύ εξειδικευμένη βιομηχανία, ε, δεν είναι εύκολο να ξαναβρούν δουλειά ε, αλλού. Δεν μιλάμε μόνο για τη Microsoft, αλλά και 8 ε, άλλες εταιρείες που είναι υπεργολάβοι ή προμηθευτές σχετικών εταιριών. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία. Το κράτος μέλος θέτει κατά μέρος υποτίθεται αρκετά κονδύλια για να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή την υποχρέωση δεν την έχει αναλάβει ε, με ε, ικανοποιητικό τρόπο το κράτος μέλος, το εκάστοτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διασφάλισαν αρκετά κονδύλια έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν έλεγχοι που θα βεβαιώσουν ότι σωστά χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα. Έχουμε επίσης και υπηρεσίες πρόσωπο με πρόσωπο για τους απολυμένους. Αυτές οι υπηρεσίες αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες. Είναι και στην περίπτωση αυτή της Microsoft ισχύει αυτό. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να προσθέσω. Δεν έχω ημερομηνίε ε, για την ε, ε, υποβολή τροπολογιών. Ενδεχομένω ο πρόεδρος μπορεί να μας μιλήσει για αυτό. Καλώ Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Για τις ημερομηνίε καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την έκθεσή σας είναι η 15η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, αυτή είναι η καταδεικτική προθεσμία για τις τροπολογίες. Η Επιτροπή για την Απασχόληση θα ψηφίσει στις 26 Σεπτεμβρίου το κείμενό σας και η δική μας Επιτροπή το ίδιο, 26-29 Σεπτεμβρίου. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο για την έκθεση του κυρίου Πέτρη Σαρβάμα. Έχετε σχόλια. Βλέπω πως όχι. Επομένως, Αυτά με αυτό το θέμα. Αναβάλλεται η έκθεση Γκονζάλες Πόντς για την Έριξον και το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Στις 15 και 50 Ακριβώς στις 15 και 50 ακριβώς πρέπει να ξεκινήσει η ψηφοφορία και είναι τώρα 15 και 50 ακριβώς. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Σας καλώ να εισάγετε την ηλεκτρονική σας κάρτα στην υποδοχή. Να κάνουμε μια δοκιμή καταρχάς για να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα δουλεύει. Άρχεται η ψηφοφορία, δοκιμαστική είναι, για να δούμε αν δουλεύει το σύστημα. Ένας δεν ψήφισε, υπάρχει κάποιος που δεν ψήφισε ενώ έβαλε την κάρτα του. Ναι, καλώς. Πέρας της ψηφοφορίας. Για την έκθεση Χριστοφόρου. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αξιολόγηση. Τροπολογία υπαριθμών 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίβεται. 17 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 19 πάλι λέει ο πρόεδρος, ο με συγχωρείτε, 20, τροπολογία 20 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 20. Πέρασε. 22 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 21. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 16 κατά. 22, η τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 24. εγκρίνεται. 25 υπέρ. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα πρέπει να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε την 25 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 17-13. 26 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Η πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 7. Πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ 16 κατά. 8 υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8η τροπολογία. περας Απορρίπτεται 21-13. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Με ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 37 υπέρ, καμία κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Προχωρούμε τώρα την έκθεση του κυρίου Αλή. Εργαλεία της κοινή αγροτικής πολιτικής για τη μείωση της μεταβλητότητας των τιμών στις, ε, αγορές γεωργικών προϊόντων. Η τροπολογία υπαριθμών 25 έχει αποσυρθεί. Λίγο πριν από τη συμβιβαστική υπαριθμών 3. 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 22 κατά 15 υπέρ. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 19 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 23 καλύπτεται από τη συμβιβαστική 1. Φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Σημαντική ψηφοφορία θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Συμβιβαστική 2 γίνεται δεκτή 25 υπέρ 12 κατά. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 31. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 20 υπέρ, 13 κατά. Δεκτή. 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 35. Ψηφίζεται. 26 υπέρ, 9 κατά. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας για να κερδίζουμε χρόνο. 36 υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτή. 37 υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ της συμβιβαστικής παρήθμου 4. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1. Ψηφίζεται. Τέλος. 20 κατά 14 υπέρ απορριφθήκε. Αυτά για την 1. Τώρα 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται, 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζεται. Τέλος. 19 υπέρ, 18 κατά. 16 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 16 ψηφίζεται. Τέλος. Η 16 επαναλαμβάνω ήταν αυτή. Τέλος της ψηφοφορίας. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται. Τέλος. 20 υπέρ 18 κατά δεκτή. Το σύνολο του τροπολογημένου πλέον κειμένου ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Τέλος. 31 υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Φτάνουμε τώρα στο τρίτο τμήμα του προϋπολογισμού 16. Κύριε Φερνάντες έχετε κάνει ορισμένες προτάσεις μεταφοράς, αν δεν υπάρχουν. Όχι, περνάμε στα άλλα τμήματα τότε. Καταρχάς, τα θέματα τα οποία δεν θα αντιμετωπιστούν και κλεισμένων των θυρών. Ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο. Θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι πράγματι ο διορθωτικός υπαριθμών 3 θα τον συζητήσουμε και κλεισμένων των θυρών. Ένα άλλο θέμα τώρα για το 4. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, Είμαι υπέρ του 4, του άρθρου δηλαδή 27 διορθώνει ο πρόεδρος. Έτσι κι αλλιώ το 27 είναι θέματα ασφαλείας που θα αντιμετωπίσουμε in κάμερα και κλεισμένων των θυρών. Για το άρθρο 25 τώρα, Μπορούμε χωρίς ψηφοφορία να κάνουμε δεκτή την πρόταση. Δεν υπάρχει θέμα. Θεωρείται δεκτό. Το λοιπόν European ούτε στο επόμενο έχουμε πρόβλημα, διακόπτει εδώ ο πρόεδρος. Πριν περάσουμε τώρα στην κεκλεισμένων των ε, θυρών συνεδρίαση, η κυρία Χολμάιερ για τα κτίρια. Αγαπητέ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία μας ε, είχε αποστείλει ένα φάκελο τον οποίο ε, να, να, να, να αναθεωρήσουμε και θα ήθελα να ξανακοιτάξω τα αριθμητικά στοιχεία τα ποσά αυτά, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, όχι μόνο μια ενημερωτική διαδικασία και το Συμβούλιο ζήτησε παραπάνω στοιχεία, γιατί τα ποσά δεν είναι σαφή και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε αυτά από την αρχή. Εγώ τα έλαβα αυτά χτες. Οι σκιώδες τα διάβασαν σήμερα μόλις, έμα ε, πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ευκαιρία να τα εξετάσουν, να, τα διαβάσουν. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να τα κοιτάξουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Καλώς, μεταφέρεται λοιπόν για την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Μια καινούργια διαδικασία να ξεκινήσει, διευκρινίζει η κυρία Ολμαϊρό, όχι να παραταθεί η προηγούμενη, γιατί χθε λάβαμε ένα καινούργιο φάκελο. Μάλιστα. Ναι, στις 14 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση ή αναθεώρηση midterm review και όχι revision. Να αντλήσουμε τα διδάγματα αυτής της διόρθωσης. Υπάρχουν άλλα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε δημόσια. Όχι. Άρα θα περάσουμε στη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Καλό όλους και όλες όσοι και όσες δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών να αποχωρήσουν από την αίθουσα.